Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής της υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ε, δίνω πρώτα το λόγο στην ε, κυρία Άστον, Baroness Άστον, the floor is yours. Uh, thank you, very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό και στην ώρα των ερωτήσεων, το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ανησυχεί ιδιαίτερα όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό τη. Οι συνάδελφοι ήδη αναφέρθηκαν ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, το, στις 23 Ιανουαρίου συζητήθηκε το θέμα της επιβολής νέων κυρώσεων. Όπως σας είπα, σε όλες τις περιπτώσεις θέλουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε τις Ιρανικές αρχές ε, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Και αυτό είναι ζωτική σημασία για την διτή αυτή προσέγγιση ε, μαζί με την ε, διαδικασία ε3-3 που όπως ξέρετε είναι η βασική διαδικασία. Είχαμε αρκετά ψηφίσματα του, ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά παρά τα ψηφίσματα η, το Ιράν εξακολουθεί να μην ε, ε τηρεί τις δεσμεύσεις, να μην ε, ακούει τι συστάσει της διεθνού Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Ξεκίνησε διαδικασίε επλουτισμού ουρανίου κατά 20% στο ΚΟΜΠ, μια στρατιωτική εγκατάσταση πυρηνικών. Όπως ξέρετε, εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες διότι δεν υπάρχει συνεργασία με το Ιράν για να λύσει αυτές τις εκκρεμότητες και ιδίω όσον αφορά τη στρατιωτική συνιστόσα του πυρηνικού του προγράμματο. Η έκθεση τη Διεθνού Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια παρουσίασε τα ευρήματά τη για τι δραστηριότητε του Ιράν για την ανάπτυξη πυρηνική τεχνολογία. Επί τη βάση αυτών, ε, το Συμβούλιο των Κυβερνητών ενέκρινε ένα ε, ψήφισμα το οποίο εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για το Ιρανικό πρόγραμμα. Τα όσα κάνουμε ελπίζω να καταδεικνύουν ότι δεσμευόμαστε για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε διπλωματική λύση για το πυρηνικό θέμα του Ιράν που είναι το δεύτερο τμήμα αυτής της διτής διαδικασίας. Εγώ μίλησα με τον εταίρο μου και καθορίσαμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκομίσει κάποια ωφέλη και στο πολιτικό και στο οικονομικό πλαίσιο. Αλλά παρά τις διάφορες υπενθυμίσεις μου δεν έχω λάβει καμία απάντηση στις προτάσεις ε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί διαδικασία εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στη βαθμιδόν προσέγγιση πάντα εκφράσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν το Ιράν, όπως για παράδειγμα τη συνεργασία σε θέματα ε, αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Και επαναλαμβάνω το ίδιο μήνυμα προς την Ιρανική πλευρά. Προσφάτως, στις συζητήσεις μου με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Σαλέη και Εκ παραλλήλου, χρησιμοποιώντα και τι επαφέ μου με τρίτε χώρε, ιδίω με την Τουρκία, προσπάθησα να διαβιβάσω το μήνυμα προ το Ιράν ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για τι διαπραγματεύσει μέσω αυτή τη διαδικασία δημιουργία εμπιστοσύνη, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή στιγμή στο Ιράν αποδείξει ότι είναι διατεθειμένο να συζητήσει επειδή ακριβώς υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία, το Συμβούλιο ενέκρινε ε, κυρώσεις και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για να επιδείξουμε ότι είναι ενωμένη η Ευρώπη και έχει ηγετικό ρόλο στα θέματα αυτά. Οι κυρώσεις ε, αφορούν τις οικονομικές δυνατότητες του Ιράν για την επιτυχία του πυρηνικού της προγράμματα ε, και, δεν, ε, και δημιουργούν προβλήματα φυσικά στα οσοδήματά τους από το πετρέλαιο και τους ορυκτούς του πόρους. Οι εξαγωγές είναι περίπου το 40% των Ιρανικών εξαγωγών και το 70% των κυβερνητικών οσόδων. Η εισαγωγή σε Ευρωπαϊκές Ένωση είναι το 20% των εξαγωγών ε, του πετρελαίου του Ιράν. Εάν λοιπόν στοχεύσουμε σε αυτή τη σημαντική ψυγή, ε, πηγή εισοδήματο, θα αυξήσουμε τι πιέσει προ την Ιρανική κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις, ε, τη μη υπαρξερνητικών αρνητικών για τον πληθυσμό του Ιράν. Οι ε, κυρώσεις των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ενισχυοί. Στις 27 Δεκεμβρίου ε, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ενισχύσουν τις κυρώσεις τους ε, και στοχεύουν κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ιράν και εισοδήματα από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών πετρελαίου. Εμείς τώρα προσπαθήσουμε να πείσουμε χώρε που έχουν την ίδια άποψη με εμά, ιδίω χώρες που εισάγουν πετρέλαιο από το Ιράν, να αναλάβουν αντίστοιχα διαβήματα και να προσπαθήσουν να περιορίσουν ε, τις εξαγωγές. Έτσι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές οι κυρώσεις. Γίνονται λοιπόν όλα αυτά ε, προσαρμοζόμενοι στην κατάσταση και προσπαθούμε να δούμε κατά πόσον έχουν αποτελέσματα τα μέτρα. Θα το εξετάσουμε αυτό στους επόμενους μήνες και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και τυχόν προβλήματα, διασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα έχουν χρόνο και μέσα να προσαρμοστούν και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει και συνέχεια στον ενεργειακό εφοδιασμό τους. Θα ήθελα τέλος να υπενθυμίσω ότι και εμεί εξακολουθούμε να ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Αυτό έχει σχέση ιδιαίτερα με τη ε, συνεχή ε, καταπίεση της αντιπολίτευσης αλλά και την ε, εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής. Επειδή αυξήθηκαν σημαντικά οι εκτελέσεις από τον, τελευταίο, από τον περασμένο Απρίλιο, Υπάρχει ένα ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα θέματα της θανατικής ποινής ε, και στοχεύει κυρίως στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, από τον Οκτώβριο και μετά ε, έχουμε 61 άτομα καταδικασμένα σε θάνατο και προσπαθούμε ε, μέσω των κυρώσεών μας να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Συνεχίζουμε να πιέζουμε προς τη ε, σωστή κατεύθυνση, πιέζουμε το Ιράν και πιέζουμε για διαπραγματεύσεις και προσβλέπω ε, στα όσα έχουν να μου πούν τα αξιότιμα μέλη για το θέμα αυτό. Άστον. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Άστον. Νομάδων. Για δύο λεπτά, ε, εκ μέρους της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Σαλαφράγκα Σάντζεθ Νέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη, εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Συμβούλιο της 23ης Ιανουαρίου πήρε μια απόφαση που ήταν δύσκολη, αλλά συνεπής. Σας συγχαίρω για αυτό κύριε Άστον και το Κοινοβουλίο θα υποστηρίξει την θέση του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου στο αυριανό μας ψήφισμα. Ήταν δύσκολο αυτό γιατί αυτό σήμαινε σημαντικέ θυσίε για πολλά κράτη-μέλη, αλλά ήταν συνεπές το αποτέλεσμα αυτό γιατί ακολουθεί τι αρχέ που έχουμε υποστηρίξει τόσο ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία, όσο και η πρωθυπουργοί της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Γαλλία, που είπαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να πάρει πυρηνικά όπλα. Πρέπει όμω να είναι αποτελεσματικά αυτά τα, μέτρα κατά του Ιράν για να επανέλθει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, να υπάρξει διάλογο, να συνεργαστεί πλήρω με του επιθεωρητές τη Διεθνού Επιτροπή Ατομική Ενέργεια και επίση κυρία Άστον για να σταματήσουν να κρούν τα τύμπανα του πολέμου. Ξέρουμε ότι ένας από τους υποψήφιους, ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ ζητά ταχεία δράση. Ξέρουμε ότι αυτές οι κυρώσεις μπορεί να είναι αναποτελεσματικές γιατί οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόνται περισσότερο το αργό πετρέλαιο από ότι το Ιράν στι ευρωπαϊκέ εξαγωγέ. Ο κίνδυνο να κλείσουν τα στενά του ορμού θα, μπορέσει να οδηγήσει, θα ίσω σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και να οξύνει και την πετρελαϊκή κρίση. Γι' αυτό, κύριε Άστον, πέραν τη εσωτερική διάσταση, πέραν τη συνεκτικότητα των θέσεων του Συμβουλίου, όπω φάνηκε και στι 23 Ιανουαρίου, είναι απαραίτητο να δράσουμε αυτή τη στιγμή και σε εξωτερική διάσταση μαζί με τους συμμάχους μας. Η θέση της Ινδίας, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε θα πετύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Η Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Μουνίθ Ντεουρκίθα. Για λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Άστον, είναι σαφές ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα του Ιράν μέσα στην, στο έτος 2012. Είναι μια χώρα η οποία οδηγεί σε περιφερειακή και παγκόσμια ακόμα αποσταθεροποίηση λόγω της έλλειψης διαφάνειας σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα και συγχρόνως επειδή είναι ένας μεγάλος εξαγωγέας αργού πετρελαίου. Ο τρίτος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι εξαγωγές του πετρελαίου είναι το 80% των εσόδων του Ιράν και επομένως είναι ευαίσθητε σε κυρώσεις. Η δική μου ομάδα, ακόμα και αν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κλιμακώσει την ένταση, η δική μου ομάδα αποκλεί την στρατιωτική επιλογή. Θέλουμε να έχουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση με τη δυτή οδό όπως αναφέρατε, δηλαδή κατάλληλε κυρώσει οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις, πολιτικούς ηγέτες και οικονομικούς φορείς για να μειωθεί η επιβολή της θέσης τους στην Ιρανική κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει να ανανεώσει και τη δεύτερη πτυχή αυτού του διτού δρόμου που είναι η διπλωματία. Θα πρέπει να επιμείνουμε να υπάρξουν αυστηρές αυστηρή έλεγχη ε, των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Ε, έγκριση από το Ιράκ όλων των μέτρων διασφάλισης που επιβάλλει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου για πολιτική χρήση όπως προβλέπει και η συνθήκη μη διασποράς των πυρηνικών όπλων. Δεν πρόκειται λοιπόν για, τον, για την κατάσταση που υπήρχε στον Οκτώβριο να πούμε στο Ιράν ότι δεν πρέπει να έχει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου σαν προϋπόθεση για το διάλογο. Όλα τα μέτρα τα οποία ζητά η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την, τον έλεγχο της παραγωγής ουρανίου θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και έτσι μονάχα μπορούν να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα δημιουργίας εμπιστοσύνης για να έχουμε καλύτερες σχέσεις με το Ιράν. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάκε για την ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, <clears throat> κύριε Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Η, ε, το Ιράν ε, εξεφράστηκε με έκπληξη για τα μέτρα αυτά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ενωμένη εις τα μέτρα που έλαβε στην απόφαση της 23ης Ιανουαρίου χρειαζόμαστε να δούμε και περισσότερα τέτοια μέτρα. Αλλά δεν είναι μοναδική μας επιτυχία να απομονώσουμε το Ιράν, αλλά να συνεργαστούμε με την Τουρκία και άλλους εταίρους κατά τρόπον ώστε να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να πείσουμε τους Ιρανούς να ξεκινήσουν μια ουσιαστική διαπραγμάτευση κατά τρόπον ώστε να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα πείσουμε το Ιράν, όχι μόνο με κυρώσεις, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μπορέσει να ανοίξει και μία εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Ιράν η οποία να μπορεί να επεμβαίνει σε περίπτωση παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διεξάγει ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Οι συντηρητικοί σε αυτό το κοινοβούλιο θεωρούν ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός σκοπός αλλά ένα μέσο για την επίτευξη ενός τόπου και θα πρέπει να υπάρξουν υπεύθυνοι οι οποίοι θα παρακολουθούν τα μέτρα τα οποία πρέπει να πλήξουν ή το πυρηνικό πρόγραμμα ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι όμως τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει συγχρόνως μία κίνηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανεξάρτητη, ιδίως σε μία χρονιά εκλογών, διότι το οι Ηνωμένε Πολιτείε επέλεξαν διαφορετικές κυρώσεις αλλά έχουν επιβάλει και έμεσες κυρώσεις μέσω των επιχειρήσεων πρέπει πάντοτε να μπορεί κανείς να στέλνει τρόφιμα και φάρμακα στο λαό του Ιράν και να έχουμε υπόψη μας τη νέα γενιά ε, και οι τεχνολογίες δεν θα πρέπει να ε, συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι δεν θα εξάγονται κατασταλτικές διαδικασίες σε αυτές τις ε, βίες χώρες οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματα. Μπλε κάρτας από τον κύριο Τάνοκ. Δέχεστε την... Ε, το ερώτημα του κύριου Τάνοκ. Η κυρία Τσάκε αναφέρθηκε σε τη συντηρητική πλευρά του Κοινοβουλίου που πιστεύει ότι οι κυρώσεις μπορεί να είναι αυτός σκοπός. Εννοεί εμάς και ε, πρέπει οι ε, κυρώσεις να έχουν πάντοτε συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Θα το πω και στην ομιλία μου αργότερα. Θα ήθελα όμως να μου πει τι εννοεί όταν αναφέρεται στη συντηρητική πλευρά του Κοινοβουλίου. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένους ευρωβουλευτές οι οποίοι πριμοδοτούν τις κυρώσεις. Το ΕΛΚ που ζήτησε χωριστή ψηφοφορία σε ένα κείμενο το οποίο θα συζητηθεί αύριο και προσπαθεί να έχει μία συνεκτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει οι κυρώσεις να πλήττουν ολόκληρο τον ε, πληθυσμό αλλά συγκεκριμένους ανθρώπους ανθρώπους μόνο και ε, ε, είπα ότι μιλώ για την συντηρητική πλευρά του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη δικιά μου πολιτική ομάδα και χαίρομαι που και εσείς θα κάνετε την ίδια διάκριση την οποία και εγώ έχω διατυπώσει. Ευχαριστώ. Ε, Κρόνμπεργκ, εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας για 3,5 λεπτά. Thank you, Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα των Πρασίνων εκφράζει τη μεγάλη της ανησυχία <clears throat> για τις εντάσεις στην περιοχή του Περσικού κόλπου και υποστηρίζει τις νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν. Ανησυχούμε όμως πάρα πολύ για το αρνητικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει για τον πληθυσμό του Ιράν. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν πάντα ότι δεν μπορούν να υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις <clears throat> για την <clears throat> διαφορά με το Ιράκ για το πυρηνικό του ε, πρόγραμμα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία και εμεί έχουμε προτείνει μια τροπολογία προ την κατεύθυνση αυτή για το ψήφισμα. Έχουμε μια διτή προσέγγιση. Έχουμε εφαρμόσει τι κυρώσει. τώρα είναι καιρό να προχωρήσουμε και σε διαπραγματεύσει. Το ερώτημα είναι πώ μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Είπε το Ιράν ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το Ιράν δεν θα διακόψει οποιαδήποτε διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου ως, προϋποθέσεις, ως προϋπόθεση διαπραγματεύσεων. Ζητούμε από όλους να συζητήσουν ειλικρινά και χωρίς προϋποθέσεις. Το Ιράν και η Δίξη έχουν διαδοχικά απορρίψει όλες τις προτάσεις για συνεργασία. Γιατί δεν υπήρξε συγχρονισμός στις προτάσεις των τριών συν των ευρωπαϊκών τριών συντριών και του Ιράν για τα θέματα αυτά διαπραγματεύσεων. Θα θέλαμε και η Τουρκία και η Βραζιλία να εμπλακούν στις διαπραγματεύσεις αυτές, γιατί είχαν ήδη προτείνει συμβαστικές λύσεις στο παρελθόν για την επίλυση αυτής της διαφοράς και θα πρέπει και πάλι να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Αν μπορέσουμε να ξανασυνεχίσουμε και πάλι τις διαπραγματεύσεις, αυτό μπορεί να ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για να φύγουν τα πυρηνικά όπλα από τη Μέση Ανατολή. Θα μπορέσουμε λοιπόν έτσι να χαράξουμε ένα καλύτερο οδικό χάρτη για αυτή την διαδικασία. Οι πράσινοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και να αποσυρθεί από την πυρηνική ενέργεια όπως έχει κάνει ήδη η Γερμανία. Το παράδειγμα του Ιράν δείχνει ότι δεν υπάρχει εύκολος, δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς την πολιτική και τη στρατιωτική χρήση των πυρηνικών τεχνολογιών πράξη καλής θέλησης που θα δείξει την διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάλογο θα πρέπει να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν και το Ιράν θα πρέπει να πάρει εγγυήσει ασφαλείας γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο μια χώρα να έρθει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όταν υπάρχει ο κίνδυνος πολέμου που επικρέμαται. Τάνοκ, εξ ονόματος της ομάδος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ε, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η φιλοδοξία ε, στρατιωτικών πυρηνικών του Ιράν και τις ε, δισταγμούς τους να τηρήσουν τις απαιτήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας δημιουργούν προβλήματα και στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή αλλά δημιουργούν και μεγάλη απειλή για την ύπαρξη του ίδιου του Ισραήλ. Επίσης ε, πλήττονται οι όμορες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και ε, οι άλλες χώρες εάν ε, το Ιράν έχει πυρηνική στρατιωτική ενέργεια θα δημιουργήσει προβλήματα στις υπόλοιπες χώρες της περιοχές. Υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία που εισάγουν ε, ε, αργό πετρέλαιο και πετρέλαιο από, την, από το Ιράν εν γέννη και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και να ε, πιεστεί το Ιράν, εάν σταματήσουν να εισάγουν πετρέλαιο, να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ε, δεν επιβάλλει τις κυρώσεις όπως ε, θα έπρεπε. Για πρώτη φορά λοιπόν μιλάμε μία φωνή και θα ήθελα να ενθαρρύνω το Ιράν να αρχίσει να τίνει ευήκονους. αντί να δείξει παράδειγμα του ένδοξου παρελθόντου τους, είναι ένα από τα θλιβερά παραδείγματα, καταπίεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εκλογές και κάνει δημοσίως ε, εκτελέσεις ομοφιλοφίλων ε, για σεξουαλικά παραπτώματα ακόμα και σε ανηλίκους και εξάγει τρομοκρατία ε, με, μέσω της Χεσμπολά στις γείτονες χώρες. Επίσης ε, παρεμβαίνει στις γείτονες χώρες όπως το Μπαχρέιν ε, ε, μέσω της δικτατορίας του. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα πρέπει λοιπόν το Ιράν να γίνει ποτέ πυρηνική δύναμη και όπως είπαν και κάποιοι άλλοι δεν θα πρέπει να υπάρξουν αποκλεισμοί σε μελλοντικέ ή περαιτέρω επιλογές να του αποτρέψουμε το να γίνει πυρηνική δύναμη το Ιράν. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία ε, εξ της Ομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, της Αριστεράς των Πρασίων, Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Frau Kollegin Ernst, Sie haben das Wort. Damen und Herren, οι πρόσφατες κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μέτρα για να ε, εξασφαλίσει κανείς και να καθησυχάσει ε, την κατάσταση. Είναι πολιτικό ε, αφελές να πιστεύει κανείς ότι μπορεί με τις κυρώσεις να λύσει το πρόβλημα διότι πρέπει το Ιράν το οποίο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 παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πρέπει να τιμωρηθεί αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέσω της, ε, ε, της διακοπής της αγοράς πετρελαίου και με αυτό δεν βοηθάμε καν και για τις εκλογές που επίκυνται στις χώρες αυτές. Αυτό πρέπει να έχετε υπόψη. Δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη εφαρμογή εφαρμογή ατομικού προγράμματος ε, ε, από το Ιράν υπάρχουν ε, υποθέσεις αλλά χρειαζόμαστε αντί για κλιμάκωση να υπάρξει διάλογος και μία ειρηνική διαβίωση και συμβίωση σε όλη την περιοχή αντί να οξύνεται όλο και περισσότερο η τωρινή κατάσταση. Ευχαριστώ. Μπέλντα Μπάστιαν, εξ της της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βρίσκεται σε μεγάλη, κάτω από μεγάλη πίεση ακόμα και η εξουσία του κυρίου, το κύρος του κυρίου Χαμένη είναι υπό συζήτηση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη διεθνή κοινότητα να μπορέσει να αποτρέψει το Ιράν από το να συνεχίσει την πυρηνική του τροχιά. Ε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξουν σοβαρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμπαγής διατλαντική κοινή θέση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Μεταβαίνει εκεί ο Αμερικανικός στόλος, υπάρχουν πολλές ε, πηγές που μιλάνε για προκλήσεις και για πόλεμο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό καθεστώς επιτήρησης από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για το Ιράν. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι λέει την αλήθεια το Ιράν και όχι να ακούσουμε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία σύγκρουση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών στη Μέση Ανατολή και αυτό εξηγεί και το γιατί το Ιράν έχει πυρηνικέ επιδιώξει. Τι θα κάνετε λοιπόν για, κάτι, για να αντιμετωπίσετε αυτή η κατάσταση. Ο κύριο Έρεν εξ ονόματο των μη εγγεγραμμένων, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι άδικο και καταπιεστικό το καθεστώς της, ε, του Ιράν και η Αυστρία, η Αυστρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, παρόλα αυτά δεν μπορεί να ζητά από το Ιράν να α, σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχει δυνητικά μονάχα ένα πυρηνικό πρόγραμμα και η έκθεση του ΟΗΕ μιλάει για απλώς ικανότητα για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια στρατιωτική ενέργεια επί τη βάση επιχειρημάτων τα οποία είναι σαθρά. Και γι' αυτό θέλω να θέσω το ερώτημά μου προς την κυρία Άστον. Ποιο είναι το σχέδιο Β σας στην περίπτωση που οι κυρώσεις δεν θα αποδώσουν τους απαραίτητους καρπούς. Τι θα πράξετε τότε. Και δεύτερον έχω να θέσω και ένα ερώτημα για το στρατόπεδο Άσουραφ. Έχει περάσει η προθεσμία για τη μεταφορά αυτού του στρατοπέδου. Υπάρχει η πρόταση τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν άσυλο σε, κρατού, σε, σε αυτούς που μένουν στο στρατόπεδο Ασράφ. Είναι μια πρόταση η οποία ακόμα είναι έγκυρη. Τι είναι, ποια είναι η άποψή σας ως ε, είπα του εκπροσώπου. Τους ε, άλλους μη εγγεγραμμένους ομιλητές. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Μπροκ, Έλμαρ Μπροκ, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι αυτά τα οποία προσπαθούμε με το σχέδιο ψηφίσματος και αυτά τα οποία ελέγχθησαν μέχρι στιγμή συνάδουν. Δηλαδή πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις, ότι οι κυρώσεις πρέπει να μην είναι αντιπαραγωγικές, να μην οδηγήσουν σε μία συσπήρωση και ε, να συνενώσουν το λαό με το καθεστώς και να αποδείξουμε ότι αυτό το καθεστώς είναι μια πραγματική δικτατορία όπου δεν σέβεται τα συμπεφωνημένα και γι' αυτό πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε περιπέτειες στα στενά του ορμούς μέσω των κυρώσεων διότι αυτές δεν είναι προς συμφέρον κανενός διότι με τις προτάσεις μας με τα, τις κυρώσεις αυτές ε, θα ενισχύσουμε ε, τους, ε, τις κινήσεις της επαναστατικής φοράς του ΡΑΝ και πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε φιλοπόλοιμοι. προσπαθούμε ανα πάσα στιγμή να αποφύγουμε τις ένοπλες σειράξεις εάν τα μηνύματα γίνουν σεβαστά και μπορεί μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις μέσω ομολόγων όπως η Τουρκία αλλά και η Ρωσία και η Κίνα οι οποίες έχουν δώσει ένα σαφές μήνυμα γενικά και θα πρέπει μέσω αυτών των μέσων να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όχι στο να σταθεροποιήσουμε ένα καθεστώς αλλά πραγματικά να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το καθεστώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των ειρηνικών πυρηνικών εφαρμογών και να μην δώσουμε σε κανέναν λαβή για να προχωρήσει σε στρατιωτικές επεμβάσεις. Ευχαριστώ. Άννα Γκόμες για δύο λεπτά. The Iranian authorities Επιμένουν οι αρχές του Ιράν να εμπλουτίζουν το ουράνιο σε ένα επίπεδο που ξεπερνάει αυτά που απαιτούνται σε ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Θέλουμε να στείλουμε σαφείς ενδείξεις σε όλους τους Ευρωπαίους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράκαμψη και πάλι των ε, κυρώσεων. Είναι πραγματικά τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί επίκυνται οι Αμερικανικές προεδρικές εκλογές και υπάρχει Πολεμοχαρή ρητορική και στι ΗΠΑ και από την πλευρά του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καταστροφή για όλη την περιοχή, ιδίω για το Ισραήλ. Στη δική μα προσέγγιση ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ευρύτερη συμφωνία με διπλωματικά μέσα, να γνωρίσουμε το ρόλο του Ιράν ω ε, περιφερειακή δύναμη και να έχουμε μια αντιπροσωπεία στην ε, περιοχή. Να περάσουμε από το καθεστώ ελέγχου των πυρηνικών όπλων σε μια παγκόσμια βάση για τα πυρηνικά όπλα που να μπορούν να ελέγχονται από όλους. Επίσης να υπάρξει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει και την ε, Σαουδική Αραβία και ενδεχομένω και το Ισραήλ για να υπάρξει το απαραβίαστο των συνόρων στην περιοχή. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και την αλληλεγγύη μας για το λαό του Ιράν που αγωνίζεται για τα βασικά του ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνουμε σαφέ ότι οι κυρώσει δεν πρέπει να έχουν το λαό του Ιράν σαν στόχο και θα έχουν αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα εάν γίνει κάτι τέτοιο γιατί απλώς θα ενισχύσουν την αντιδυτική προπαγάνδα του καθεστώτος στο Ιράν. Αλεξάνδερ Γκραφ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχω και εγώ εκφράσει την ικανοποίησή μου για την απόφαση του Συμβουλίου να εφαρμόσει κυρώσεις για το Ιράν. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι και σωστό και πρέπει. Αλλά πολλοί συνάδελφοι είπαν εδώ ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις στρατιωτικές ε, προθέσεις του Ιράν και δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει τα στρατιωτικά από τα, πολιτικά προγράμματα. 5.000 κιλά, κιλά ουρανίου εμπλουτισμένο στο 3% αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ε, επαρκές για μια πολιτική χρήση, αλλά 500 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένο στα 20% αυτό μόνο για στρατιωτικούς σκόπους μπορεί, σκόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και αυτά είναι σαφή από την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ότι υπάρχει πρόθεση χρήσης της ποινική ενέργειας για, τους, για στρατιωτικούς στόχους. Γι' αυτό είναι απόλυτα σωστό να ασκήσει μεγάλη πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα εκτοξεύσεως ποινικών κεφαλών. Τους ε, πυράβλους του οι οποίοι όλο και περισσότερο εξελίσσονται από το Ιράν. Επομένως πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν η εφαρμογή του εμπάργου για την παράδοση πετρελαίου με την ε, προσπάθεια όλων των κρατών μελών να βρουν εναλλακτικές λύσεις από την τροφοδοσία για το Ιράν. Πιστεύω ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ευρεία υποστήριξη και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τον θετικό και επικοδοματικό ρόλο της ε, Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με τον νέο διευθυντή της και πιστεύω ότι μπορεί και η Τουρκία να παίξει ένα σημαντικά επικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα μαθήματα της Αραβικής ε, Άνοιξης ισχύουν και για το Ιράν, όπως και για οποιαδήποτε άλλη καταπιεστική κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο. Ο Αχμαντίνετζάν και οι φασίστες συνάδελφοί του στο Ιράν ε, δεν είναι αλόβητοι στον ε, άνεμο της αλλαγής που πνέει στην ε, Αραβική Χερσόνησο. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό όπλο για να επιβάλλουν εκ νέου την εξουσία τους στην περιοχή και να εκβιάσουν όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζουμε λοιπόν την αποτυχία της πολιτικής μας που προσπαθεί να τους κατευνάσει. Προσπαθεί, ε, ε, η πολιτική αυτή ουσιαστικά τους έδωσε περισσότερο χρόνο για να παράξουν περισσότερη τρομοκρατία παγκοσμίων και να κατασκευάσουν πυρηλικά όπλα στη χώρα τους, ε, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταπιέζουν το λαό. Αυτό λοιπόν το πυρηνικό τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν είναι μία από τις λίγες χώρες που εξακολουθεί να υποστηρίζει τον Ασάντ στη Συρία. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου με αυτούς του τυράννους, να προσπαθήσουμε λοιπόν να αλλάξει το καθεστώς. Τα ατομικά όπλα είναι τα τρομερότερα όπλα τα οποία υπάρχουν και θα έπρεπε να καταργηθούν διεθνώς και δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την πολιτική χρήση της ατομικής ενεργείας. Γι' αυτό και πρέπει να ταχθούμε κατά της χρήσης ατομικής ενεργείας και να υπάρχει μία ζώνη ειρηνική αφοπλισμού από ατομικά όπλα ή στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Αλλά μέχρι στιγμής το Ιράν έχει υπογράψει την ε, συμφωνία για την ε, μη διάδοση των πυρνικών μέτρων και ε, σε αντίθεση με την Ινδία και άλλες χώρες και άρα μπορεί να έχει απαιτήσει, πράγμα το οποίο είναι επικίνδυνο όπως είναι επικίνδυνο και για άλλες χώρες αλλά κανείς δεν έχει την ε, ιδέα να ε, επιτεθεί κατά οποιασδήποτε χώρας έχει ατομικά εργοστάσια. Δεν υπάρχουν λοιπόν αποτελε... αποδείξεις ότι ε, στο Ιράν ε, χτίζονται ή εξελίσσονται ε, τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχει μία πολύ δραστική κατάσταση η οποία εντείνει τον βιομηχανικό πόλεμο και ε, συσπυρώνει το Ιράν και βλέπουμε ότι ε, τα, ε, η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα για μία ακόμη φορά θα πέσουν στο βωμό των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διαδικασία της μπλε κάρτας. Δέχεστε κυρία, δέχεστε κυρία Λόζινγκ. Δέχεστε ε, κυρία Λιόζινγκ. Erlauben ε, Μπενζή. Frau Just one more time, please. I did not hear you. Yeah, ο κύριος Μπέλτα ε, επικαλείται τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Δέχεστε την, την ερώτηση του κυρίου Μπέλτα. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Κύριε Μπέλτα. Κύριε ε, κυρία Λέζινγκ, έχω μία ερώτηση. Γνωρίζετε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επανειλημμένως ε, έχει απειλήσει με εξαφάνιση το Ιουδαϊκό κράτος του, του Ισραήλ. Ε, οπότε θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αντίδρασή σας σε αυτό. Θα χρησιμοποιούσατε τις ίδιες μεθόδους. Προφανώς το γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζω τι σχέση έχει αυτό το θέμα με την ερώτησή σας. Προβέρα. Για ένα λεπτό. Grazie, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι Άστον, είναι δύσκολο να είναι κάποιος αισιόδοξο. Η διαδικασία πυρηνικών όπλων από πλευρά Ιράν θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή μεταξύ της Μεσογείου και του Καυκάσου και μπορεί να ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου πυρονικών εξοπλισμών στις ε, γείτονες χώρες ε, που μπορεί να φοβούνται το Ιράν, όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αριβία ή η Τουρκία. Υπάρχουν ε, όπλα τελευταίας γενεά, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία και θα μπορούσαν ε, να δώσουν τη δυνατότητα στο Ιράν να απειλήσει, να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ. Ένα ε, πυρηνικό ε, στρατιωτικό Ιράν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στα στενά του Ορμούς και να δημιουργήσει στρατιωτικά και πολιτικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λοιπόν μια νέα Βόρεια Κορέα στη Μέση Ανατολή. Οι νέε κυρώσει που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφώ θετικέ, αλλά πιέζει ο χρόνο και πρέπει να εξεύρουμε μια διπλωματική λύση για την κρίση αυτή και να αποφύγουμε τη στρατιωτική στρατιωτική επιλογή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ομπαμάια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει αποφασιστεί η διακοπή της τροφοδοσίας σε πετρέλαιο και πρέπει όλες οι χώρες αυτές οι οποίες τροφοδοτούνται με πετρέλαιο να σταματήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο μέσα στα πλαίσια τις ε, συμφωνίες των κρατών μελών. Θα πρέπει όμως να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάσταση των πολιτών, των απλών πολιτών στο, στο, στις χώρες αυτές οι οποίες ε, τροφοδοτούνται με, το, με πετρέλαιο από το Ιράν αλλά και των πολιτών του Ιράν οι οποίοι θα πληγούν από, από αυτό το εμπάργο. Αυτό θα επιτύχει ακριβώς τους αντίστοιχους τους αντίθετους, το αντίθετο αποτέλεσμα και υπάρχουν πολλοί εξόριστοι από το Ιράν που μας προειδοποιούν ότι θα επιτευχθεί ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν, δεν πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε τέτοια αντιπαραγωγικά μέτρα και δεν πρέπει να προχωρήσει σε κλιμάκωση της κρίσης και της έντασης. Ο κύριος Πρέντα, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την ομάδα του ΕΛ και να αποφασίσει να επιβάλλει κυράσει ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, Ιράκ είναι, στο Ιράν συγγνώμη, είναι σίγουρα θετική απόφαση. Μετά από ε, το πάγωμα πολλών επιχειρήσεων μετά από τον περιορισμό των εξαγωγών ευαίσθητων περιοχών και επενδύσεων στον τομέα των ε, πετρελαίου ε, του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων ε, το επόμενο βήμα ήταν αυτές οι κυρώσεις ε, που είναι πολύ σημαντικές για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. Ε, όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται ελαφρά την καρδία. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν αυτά τα μέτρα διότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, της πυρηνικής ανάπτυξης ε, του προγράμματο του Ιράν και μα ανησυχεί όλο και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πολύ σημαντικέ αυτέ οι κυρώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι μπορεί να εμείνει στι θέσει τη και η σταθερότητά μας και η σαφή μα θέση δίνει ένα μήνυμα προ του Ιρανού ότι δεν θα δεχτούμε στο μέλλον αυτή την απειλή του πυρηνικού στρατιωτικού προγράμματος. Ε, όσοι θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν αποτελέσματα, θα ήθελα να πω δύο σημαντικά πράγματα. Καταρχά, οι κυρώσει σίγουρα ε, δημιουργούν πρόσκομα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν επιτρέπουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Επίση, ε, το Ιράν. Ε, το ίδιο ε, διαπιστώνει ότι τα μέτρα αυτά έχουν επιπτώσεις για την οικονομία του και έτσι θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Uh, Mr. Fox. Uh, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ο κύριος Φόξ ε, ε, θέλει να κάνει ερώτηση κάνοντας χρήση της μπλε κάρτας. Το αποδέχεστε? Please, Mr. Fox. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα συμφωνεί μαζί μας ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στη Μέσο Ανατολή ε, είναι ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα συμμορφωθούν με τις επιταγές της διεθνούς κοινότητας. Ε, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ομιλήτρια είναι η κυρία Κάθλιν ε, Φανμπρέμπτ. Για δύο λεπτά. Um, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον, πέραν των παραταξιακών θέσεων υπάρχει μια ευρεία συνένεση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η επιμονή της Ιρανική κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και μα έχει υποχρεώσει να περάσουμε σε κυρώσει. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονε σε αυτήν την αίθουσα. Εγώ έχω βέβαια κάποιε ανησυχίε, γιατί υπάρχουν πολλέ περιπτώσει όπου τα, οι κυρώσει έχουν οδηγήσει μεν σε αλλαγή καθεστώτο. πρέπει όμως να είμαστε και επικριτικοί για τις κυρώσεις και το αποτέλεσμά τους εν γέννη. Η ομάδα μου και εγώ η ίδια θεωρούμε ότι αυτές οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να είναι η απαρχή μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια ένοπλη σύραξη ή μια στρατιωτική επέμβαση στην, στο Ιράν στην περιοχή. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει η στρατιωτική απειλή για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουμε ακουστοί μια στρατιωτική σύραξη θα είναι αρνητική και για το Ιράν αλλά και για την Ευρώπη και δεν πρέπει να ανέβει στις επιλογές μας. Δεύτερον, <clears throat> σε ευρύτερο πλαίσιο, το είπε η κυρία Άστον ήδη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση των πολιτών του Ιράν και τα δικαιώματά τους. Και εδώ ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες πουλάνε τεχνολογία, εξάγουν στο Ιράν τεχνολογία που βοηθάει για να υπάρξει καταστολή του πληθυσμού. Τεχνολογίες, παραδείγματος χάρη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών ή φιλτραρίσματος του ίντερνετ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι πρώτα εμείς θα κοιτάξουμε και τη δική μας ενοχή στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ακολουθεί. Κυρία Παρβάνοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, είπατε εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση στο Ιράν αποδεικνύει όλο και περισσότερο ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσω το πρόβλημα από πλευρά διεθνού κοινότητα. Δεν θα πρέπει δεν να ξεχνούμε και θέματα τα οποία είναι συνεχώ στο προσκήνιο, όπω για παράδειγμα η κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομική ενέργεια ιδίως ε, την ε, πιθανή πολιτική διάσταση του πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να η πρόσβαση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε όλες τις εγκαταστάσεις όπως ζητά η υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ρεαλιστική και ευθεία προσέγγιση για τι κυρώσει του Ιράν. Κύριε εκπρόσωπε, Εάν οι κυρώσεις δεν έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, πώς μπορείτε να μας πείτε ότι ε, σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και με την Τουρκία για να μπορέσουμε να έχουμε μια εφικτή λύση και πόσο είναι αφικτός ένας διάλογος απευθείας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Νίκη Τζαβέλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, παρακαλώ θερμά προσπαθήστε διπλωματικά ακόμα. Δεν είμαι σίγουρη ότι η δυτική διπλωματία έχει τον πρέποντα τρόπο προσέγγισης προς το Ιράν. Χρειάζονται σεβασμό, έχουν μια ιστορία 4.000 ετών, θα πρέπει να ανταλαμβάνουμε υπόψη. Τρία σημεία. Πρώτον, υπάρχει μια λεπτή γραμμή όταν βάζουμε κυρώσεις. Ποιος επηρεάζεται περισσότερο, η ελίτ η οποία κυβερνά ή ο λαός φοβάμαι ότι είναι ο λαός ο οποίος θα πληγεί, θα πληγεί σε αυτή την περίπτωση και θα έχουμε ένα μπούμεραν. Το δεύτερο είναι κυρώσεις επί της ενέργειας. Ενέργεια σημαίνει συμβόλαια πολυετή, 40 και 50 χρόνια, υποδομές μεγάλες, σημαίνει αύξηση των ειδών κατανάλωσης σε όλο τον πλανήτη. Είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά και να προχωρούμε με μια διαδικασία η οποία μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Προσπαθήστε διπλωματικά παρακαλώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τζαβέλα. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ντάιαν Ντότζ. Για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είπατε εκπρόσωπε. Είναι σωστό το να ανησυχούν οι κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για την απειλή στην παγκόσμια ασφάλεια που προκύπτει από το πρόγραμμα αυτό. Όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, είναι ένα ασταθέ καθεστώ, ένα βίαιο, συγγνώμη, ομό καθεστώ, το οποίο, το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την κατάσταση των ε, πολιτών του και επίση και η στάση του Ισραήλ κάνει τη Μέση Ανατολή να είναι πυρητή αποθήκη. Είναι απαραίτητο όμω να υπάρξουν σωστέ κυρώσει ώστε να ενθαρρυνθεί το Ιράν να μπει σε διαπραγματεύσει με τη διεθνή κοινότητα. Περαιτέρω ε, κλιμάκωση του πυρηνικού προγράμματο που οδηγεί φυσικά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλε ενέργειε οι οποίε θα οδηγήσουν στο κλείσιμο των στενών του ορμού θα είναι απόλυτα απαράδεκτε. Χαιρετίζω τη στάση τη διεθνού κοινότητα για τα θέματα αυτά. Η στάση όμω των Γάλλων και των Άγγλων που στείλανε και των Αμερικάνων που στείλανε στρατιωτικά, ε, μάλλον πολεμικά πλοία στην περιοχή αυτή δίνουν το σωστό μήνυμα. Πρέπει όλοι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίσουν το διάλογο και τη διπλωματία. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το ατού και να το υποστηρίξουμε με την απειλή ενδεχόμενης δράσης εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί. για Κύριε Πρόεδρε, Βαρόνι Άστον, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μία νέα και δύσκολη φάση των σχέσεών μας με το Ιράν ή μάλλον στην έλλειψη σχέσεών μας με το Ιράν και η ε, έκθεση της, του Οργανισμού Πυρηνικής Ενεργείας επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει και τη βούληση και τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πράγμα το οποίο η χώρα έχει κρύψει μέχρι στιγμής και από τους επιθεωρητές οι οποίοι βρίσκονται εκεί και τώρα. Διεθνώς ε, το Ιράν μας έχει απειλήσει ε, να, ότι θα κλείσει τα στενά του ορμούς και ότι θα στραφεί προς ε, τους συμμάχους μας. Έχουμε διάφορες ανησυχίες και δεν πιστεύουμε ότι ότι οι εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο θα αλλάξουν την πολιτική της χώρας αυτής. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία μοναδική λύση δηλαδή ε, να επιβάλλει κυρώσεις και ε, να διευκρινίσει στο Ιράν ότι δεν μπορούμε πλέον να στηρίξουμε αυτό το αντιδημοκρατικό καθεστώς αγοράζοντας το πετρέλαιό τους. Τώρα λοιπόν πρέπει να πιέσουμε το Ιράν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν ε, μπορεί ε, να είναι απλώς για το Θεαθήνε και για να κερδίσει κανείς ε, χρόνο και να τους επιτρέψει να αναπτύξουν περισσότερο το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Κυρία δεν πρέπει να δεχτείτε τίποτα λιγότερο από μία πραγματευτή διαπραγμάτευση και ανταλλαγή από απόψεων. Μπορούμε να δεχθούμε ε, την ε, ανανέωση της ε, ανανέωσης συμφωνίας πόρων από το Ιράν εφόσον το Ιράν σεβαστεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τη συνθήκη της μης αποδοχής πυρνικών όπλων. Μαρία Ελένη Κοπά για δύο λεπτά. Κύριε Κοπά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέδη Άστον, η σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγάλη σημασία. Η επιβολή των νέων κυρώσεων κατά τη Τεχεράνη ήταν απολύτω επιβεβλημένη. Εξίσου όμω επιβεβλημένη είναι και η προσπάθεια να εξαντλήσουμε όλε τι δυνατότητε έτσι ώστε το Ιράν να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τι κυρώσει, αν και αναγκαία, δεν είναι απλή εκτός του, ότι θα έχει ως συνέπεια να αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου παράλληλα δημιουργεί πρόβλημα στα ενεργειακά αποθέματα πολλών χωρών. το οικονομικό κόστος εξάλλου ειδικά για τις χώρες του νότου λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική κρίση θα είναι μεγάλο. από την άλλη μην ξεχνάμε ότι το ιράν έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει το πετρέλαιό του σε άλλες αγορές πέραν των ευρωπαϊκών. υπάρχει όμως και κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις θα είναι απόλυτα στοχευμένες και θα πλήξουν όσο το δυνατόν λιγότερα τον ιρανικό λαό. θεωρώ ε, λέει άστον ότι θα πρέπει να εξαντλήσετε όλα τα μέσα έτσι ώστε να πιστεί το ιράν να συνεργαστεί επικοδομητικά στο πυρηνικό ζήτημα. αλλά δεν πρέπει να είναι το μόνο ζήτημα. η διεθνής κοινότητα και η ευρώπη δείχνει να έχει ξεχάσει τη φρικτή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. νομίζω ότι πρέπει ξανά να θυμίσετε την τεχεράνη να του ευαισθητοποιήσετε ξανά για αυτό το θέμα. σε κάθε περίπτωση πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευθεί η ένοπλη σύραξη. δεν συμφέρει κανέναν μια σύραξη στην ήδη επιβαρημένη περιοχή του αραβικού κόσμου. η κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι ηνωμένε πολιτείε σχετικά με το κλείσιμο των στενών του ορμούζ φοβάμαι ότι κλιμακώνει επικίνδυνα την κατάσταση όμως το ιράν πρέπει να πείσει έμπρακτα τη δύση για την ειρηνική χρήση του πυρηνικού της προγράμματος αλλά και τη διάθεση να συνεργαστεί και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κοπά. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νίκ Γκρίφιν. Για ένα λεπτό. Τα όπλα μαζικής καταστροφής οι πολιτικοί μας ετοιμάζονται τώρα να ζητήσουν δράση κατά του Ιράν γιατί έχει όπλα μαζικής καταστροφής. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει στο παρελθόν και το ίδιο πράγμα, το ίδιο ψέμα χρησιμοποιείται τώρα για να δικαιολογήσει ένα πόλεμο κατά του Ιράν. Μπορεί να ήταν καλέ οι προθέσει στην περίπτωση του Ιράκ, αλλά εκατοντάδε χιλιάδων παιδιών στο Ιράκ πέθανε γιατί δεν είχαν τροφή και φάρμακα. Τώρα μιλάμε για πυρηνικά όπλα ε, καταστροφής στο Ιράν. Αλλά τα θύματα θα είναι πάλι τα παιδιά στο Ιράν. Γιατί ένα επιτυχές εμπάργο στο πετρέλαιο δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να έχει τροφή και φάρμακα για τον πληθυσμό του. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τέτοιες κυρώσεις, δείχνει ότι είναι χρεοκοπημένη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ηθικά. Αν οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να κάνουν πόλεμο με το Ιράν ή το Ισραήλ, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Εμεί πρέπει να μείνουμε έξω από κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω αν είσαστε έτοιμος να δεχτείτε μια μπλε κάρτα, αλλά θέλω να χαιρετήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που είναι παρόντα και να σας πω ότι πρώτη φορά που προεδρεύω, στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω και τη μητρική μου γλώσσα. Transfer for a blue card. Σε την μπλε κάρτα. Ο κύριος Τάνοκ. Ο κύριος Γκρίφιν έχει μια αδυναμία με το Ιράν για τις, ε, τις ε, του κατά του Ισραήλ. Νομίζω ότι εκεί που έρχεται το κόμμα του πράγματι το καταλαβαίνει αυτό. Ένα πιο σοβαρό ερώτημα όμως θέλω να του θέσω. Αν πιστεύει ότι το Ιράν ακολουθεί ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, τότε γιατί χρειάζεται ουράνιο ε, εμπλουτισμένο με 20 ή ακόμα και 50%. 30 δευτερόλεπτα κύριε Γκρίφιν. Δεν είμαι φίλος του Ιράν. Είμαι επικριτής του Ισλάμ και όλων των Ισλαμικών απειλών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για τη Μέση Ανατολή είναι υπόθεση των χωρών της Μέση Ανατολής. Δεν είναι δικό μας θέμα να παρέμβουμε. Αν δουν οι Ιρανοί τι έγινε στη, Λιβύη, στη Λιβύη που δεν είχε όπλα μαζικής καταστροφής, τότε δεν μπορεί κανείς να περιμένει να μην υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Έχουμε ακούσει όμως τα ψέματα για τα όπλα μαζικής καταστροφής στο παρελθόν και τώρα μάλλον τα ξανακούμε. Ο κύριος Σέφλιν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν ε, να σας ε, ε, συγχαρώ και θα συνεχίσω αγγλικά. Το πρόγραμμα του Ιράν είναι διαφυσβήτητα μία πηγή κινδύνου για όλη την περιοχή της Ευρώπης και της Ασίας αλλά δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το θέμα διότι μπορεί να μας διαφύγουν άλλες στρατηγικές εξελίξεις διότι το Ιράν στρατιωτικά δεν χρειάζεται τα πυρηνικά όπλα μπορεί να κλείσει τα στενά του ορμούς και αυτό ανεφέρθη ήδη πράγμα το οποίο θα επηρεάσει όλες τις εξαγωγές από όλο την περιοχή του Περσικού κόλπου και θα επηρεάσει και την κατανάλωση. Εάν λοιπόν το Ιράκ γίνει δορυφόρος του Ιράν τότε ε, θα έχουμε προβλήματα ε, και οι εξεγέρσεις εις το Ιράκ θα επιδεινώσουν την κατάσταση υπάρχει και ε, το καθεστώς του Ασάντ και χρειάζεται τότε και τότε θα επιτευχθεί ο στόχος του, Ιράκ, του Ιράν που είναι να κλείσει τα στενά του ορμούς, να αποκλείσει πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και να πετύχει τους στόχους του. Ευχαριστώ. για δύο λεπτά ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, πρόκειται για μια πολύ σημαντική περιοχή όπου αποφασίζουμε εάν μπορεί να αναπτυχθεί το μέλλον μας ειρηνικά και εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα διότι τώρα ε, θα πρέπει να εξελιχθεί μια κατάσταση η οποία ε, έχει διάφορες παραμέτρους και επανειλημμένως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να ε, προειδοποιήσει το Ιράν το οποίο ε, αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις και ε, κοροϊδεύε όλες τις προσπάθειες που έγιναν για διπλωματική λύση. Χρειάζεται λοιπόν μία συνεκτική πολιτική κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το καρότο και το δεί, ε, Μια με το καλό και μια με το κακό. Πρέπει όμως ε, ήδη να ε, σκεφτούμε ότι το καλό θα πρέπει να γίνει πιο προφανές κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία πίεση για το καθεστώς στο Ιράν και για να μπορέσει να υπάρχει συνεκτικότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Να αποφύγουμε η διαμάχη αυτή να οδηγήσει σε μία ένοπλη σύραξη διότι έχουμε δυστυχώς πολλά τέτοια παραδείγματα σε, αυτό, σε αυτή την Ήπερο και ε, ο πόλεμος θα ήταν καταστροφικός για το λαό του Ιράν θα, και ενέπλεκε και το Ισραήλ και θα μας πήγαινε πίσω δεκαετίας. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να απευθυνθεί μία ένοπλη σύραξη στην ε, οποία θα καταλήξουμε εάν δεν δοθεί μία μια ειρηνική απάντηση. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αντρική Ενέ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει εμπάργκο στις εισαγωγές πετρελαίου, να μην έχει νέες συμβάσεις, να παγώσει τα εισοδήματα του Ιράν από το πετρέλαιο και μαζί με τα μέτρα των ήπα ε, θα μπορέσουν να επιβάλλουν σημαντικές κυρώσεις, όπως είπε και η Υπουργό Εξωτερικών η Χίλαρη Κλίντον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν. Και είναι ε, πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίε εμπλέκονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πιστεύω ότι οι κυρώσει θα επιτύχουν το στόχο του. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα κάτι μελη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν ποιε είναι οι ενδεχόμενε συνέπειε και να είναι έτοιμε να τι ε, αντιμετωπίσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του κάνει μια στεναρή δήλωση ότι υποστηρίζει την ε, δυτή προσέγγιση και κυρώσει και διαπραγματεύσει προ το Ιράκ. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι να τονίσουμε στο Ιράν ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε το Ιράν να μείνει σε επίπεδο μιας χώρας όπως είναι η Ιαπωνία που έχει την πυρηνική ικανότητα αλλά έχει αποφασίσει να μην έχει πυρηνικά όπλα. Και κλείνω. Αυτό που θα μπορούσε να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις είναι οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στο Ιράν και ιδίως η δημοκρατικοποίηση μέσα Μέση Ανατολής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος Κουτάς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ιράν βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή τα ιρανικά πυρηνικά όπλα αποτελούν έναν επιπλέον κίνδυνο για την ειρήνη της περιοχής. Είναι μια μέθοδος για να ασκηθεί έλεγχος ε, στις ε, γείτονες χώρες και πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις προθέσεις της συγκεκριμένη χώρας. Ωστόσο, θα πρέπει να θέσουμε και το εξής ερωτηματικό. Γενικευμένες κυρώσεις για το Ιρανικό Πρετρέλαιο είναι αυτές οι οποίες θα μας οδηγήσουν ε, στην κατάλληλη λύση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πλήξουμε μια ολόκληρη κοινωνία για τα σφάλματα τα οποία ε, διαπράττει η άρχουσα τάξη. Θα πρέπει λοιπόν οι κυρώσει να ε, στρέφονται προ αυτού που κρατούν την εξουσία. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή τη κυρία Άστον στο γεγονό ότι θα πρέπει να αξιολογούμε συνεχώ τι επιπτώσει αυτών των κυρώσεων. Εκ παραλλήλου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει συνεχώς το διάλογο με την Ιρανική πλευρά. Και όπως ακούστηκε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ε, σχέσεις που έχουμε και που έχουν οι Ιρανοί με την Τουρκία. Δεν θα πρέπει δεν να λησμονούμε ότι υπάρχει το, και τα, θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι μόνο το πυρηνικό πρόβλημα όπως υπονθύμησαν πολλοί συνάδελφοι. Για αυτή την τελευταία πτυχή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει από τις ε, ε, επιχειρήσεις της ε, να επιτύχει ε, πάυση των εξαγωγών των προϊόντων ε, τους κυρίως τα ηλεκτρονικά προϊόντα έχω κατά νου και να πω ότι η μόνη λύση στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν με το Ιράν θα είναι η ειρηνική λύση. Η στρατιωτική παρέμβαση θα είναι μοιραίο σφάλμα το οποίο θα δημιουργήσει και καταστρεπτικές συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στην ε, παρέμβαση της ΥΠΑ εκπροσώπου θα πρέπει να πει ότι είναι αντίθετη σε μια στρατιωτική παρέμβαση και θα πρέπει να δηλώσει ανοιχτή για διάλογο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάτσμαρεκ από την ομάδα του ΕΛΚ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει θέση για το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η, Ευρωπα... η Παγκόσμια Υπηρεσία ε, Πυρηνικής Ενέργειας έχει εκφράσει πάρα πολλές ανησυχίες για την ενδεχόμενη στρατιωτική χρήση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Υπάρχουν και αποδείξεις ότι κινείται προς την κατεύθυνση αυτό το Ιράν. Όλα αυτά όμως δεν έχει, έχουν οδηγήσει το Ιράν να συμμορφωθεί με το καθήκον του κάτω από τη συνθήκη μη διασποράς των πυρηνικών όπλων και την υποχρέωσή του να ανακοινώσει τις ε, ενέργειες που κάνει σε πυρηνικό επίπεδο. Το Ιράν λοιπόν δεν έχει δεχθεί την, ε, και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις, ε, και τις προτάσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Πυρηνικής ε, Ατομικής Ενέργειας. Αυτή τη στιγμή αποτελεί λοιπόν μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή η κυβέρνηση του Ιράν. Θα ήθελα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο αυτό να μην ξεχάσουμε και την κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο Αστράφ. Αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την επίλυση αυτού του προβλήματο με κοινέ ενέργειε. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Σα ευχαριστώ για το γεγονό ότι παραμείνετε μέσα στο χρόνο σα. Ο κύριο Στάσιν έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι, ε, Ιρανοί πρόσφυγες μεταφέρθησαν σε ένα άλλο στρατόπεδο που μοιάζει με στρατόπεδο φυλακής και το, αυτή η μετακίνηση στο στρατόπεδο Αστράφ έγινε χωρίς να υπάρχει συνένεση ε, του Προέδρου και θα πρέπει κυρία Άστον και Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν πιο ενεργή εφόσον ε, δεν ε, υπάρχει ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις διότι υπάρχουν πολλοί φυλακισμένοι που έχουν σχέση με την Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους και να μπορέσουμε να ε, συμβάλλουμε στην επίλυση της καταστάσεως. Είναι δε ο κύριος Ελμπασράφη καλύτερη μας ελπίδα για για μια, ένα δημοκρατικό Ιράν. Ευχαριστώ. Ε, κερδίσατε και χρόνο και σας ευχαριστώ. Και ο τελευταίος εις τον κατάλογό μου ο κύριος Φέλνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι οι κυρώσεις ε, οι οποίες έχουν διατυπωθεί θα πρέπει να τύχουν της πλήρης ε, στήριξής μας είναι ένα διαφορετικό θέμα αλλά πιστεύω ότι έχουν τύχει ευρείας στήριξη ε, στην Ευρώπη και δεν νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι μία έλλειψη επιτυχίας αλλά αντιθέτως ότι αποδίδουν οι κυρώσεις που διατυπώθησαν και στηρίζουν την αντιπολίτευση στο Ιράν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ε, αυστηροί απέναντι στο Ιράν, να μην πληγεί ε, ο λαός και ε, να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση από τη διεθνή κοινότητα η οποία θα έχει ένα κόστος αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι εννοούμε αυτά τα οποία λέμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ τώρα. Λέμε πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχει ενιαία φωνή στα θέματα του εξωτερικών σχέσεων. Τα κράτη-μέλη όμως τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της διακοπής, ε, της ενδεχόμενης διακοπής ε, παροχής πετρελαίου από το Ιράν, παρόλα αυτά κατάφεραν να συμφωνήσουν με τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Οι δηλώσεις της κυβέρνησης του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένες και δεν είναι πιστικές. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παραμείνει στεναρή και θα καθορίσει το αν θα υπάρξουν και περαιτέρω κυρώσεις στην οικονομία του Ιράν. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να εξαλείψουμε τις απειλές για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Είναι κρίμα που κάποιες χώρες που έχουν περιφερειακές φιλοδοξίες δεν καταφέρνουν να ακολουθήσουν την ίδια οδό όπως και άλλες χώρες. Και αναφέρομαι στη Ρωσία και δεν βοηθούν τη διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία για ένα λεπτό. Παρβάνοβα. Ευχαριστώ για το λόγο που μου δίνετε. Είναι εντυπωσιακό το ότι το Ιράν εξακολουθεί να μην τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του αν θέλουμε να, σε, να υπάρξει σεβασμός σε αυτές τις υποχρεώσεις, αν θέλουμε όλα αυτά να σημαίνουν κάτι, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας. Γι' αυτό υπογραμμίζουμε πλήρως την ανάγκη να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί του Ιράν. Είναι απαραίτητο όμως να τονίσουμε ότι αυτές οι κυρώσει θα πρέπει να έχουν σαν στόχο το καθεστώς του Ιράν και όχι τους απλούς πολίτες του Ιράν, που είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη ζωή τους. <clears throat> Πέραν τούτου, Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση, η οποία είναι η διπλωματική διάσταση, η διάσταση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Είμαι πεπισμένη ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε να πείσουμε το Ιράν ότι πράγματι μας ενδιαφέρει να έχουμε μια σωστή σχέση με χώρες όπως το Ιράν, όχι την ηγεσία αλλά την ίδια τη χώρα, τότε μπορούμε να πετύχουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα αναχαιτήσουμε και την διάδοση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Αγκουράκη. Κύριε Πρόεδρε, η επιβολή εμπάργου στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και οι άλλες κυρώσεις που ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο αποτελούν επιθετικές ενέργειες και κλιμάκωση των μέτρων σε βάρος του λαού του Ιράν. Τα μέτρα θα εκτινάξουν τις τιμέ των καυσίμων και τα κέρδη των πολυεθνικών, θα οξύνουν ακόμα περισσότερο την καπιταλιστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγορεύεται ξανά σε παγκόσμιο χωροφύλακα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό υπαγορεύουν οι υπεριαλιστικέ αξίε και τα συμφέροντά τη. Αυτό επιβάλλει ο ανταγωνισμό με άλλε δυνάμει στο Περσικό κόλπο και στην Κεντρική Ασία. Αποτελεί πρόκληση ο εκβιασμό που επιχειρούν οι πυρηνικέ δυνάμει με πρόσχημα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι οι ίδιε αυτέ οι δυνάμει που καλύπτουν την επιθετική πολιτική και τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ, τα αμέτρητα πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη και τη διάδοση των πυρηνικών στην Ινδία και Πακιστάν. Είμαι βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι θα καταδικάσουν τι προκλητικέ αυτέ ενέργειε. Πρέπει να ματαιώσουν τα κοινά γυμνάσια ορισμένων χωρών με το Ισραήλ και τον πόλεμο σε βάρο του λαού του Ιράν. Σήμερα είναι επίγουσα ανάγκη η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια λαϊκή εξουσία έτσι ώστε οι λαοί να μην πληρώσουν με το αίμα του υπεραλιστικού πολέμου. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Είστε διατεθειμένος να απαντήσετε. Δέχεται ο κύριος Αγκυράκης. Παρακαλώ κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι βαρέθηκα να συγκρίνεται η ειρηνική αναζήτηση πυρηνικών όπλων στα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ, στο Πακιστάν ε, και την Ινδία η, Ιραν, η, το, Ινδία δεν έχει προσυπογράψει την ε, Συμφωνία Μη Διασπειράς Πυρηνικών Ιουπλών. Το Ιράν το έχει κάνει. Ο κύριος Αγκουράκης αναφέρεται ε, στο χωροφύλακα παγκοσμίω. Ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι χωροφύλακα, είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια. Πού είναι το κακό λοιπόν, γιατί το Ιράν να μην υποχρεούται να τηρήσει τις διεθνούς του υποχρεώσεις, κύριε Αγκουράκη. Μπορείτε να απαντήσετε. Καταρχήν δεν αναφέρθηκα, ε, δεν αφορούσε τα όσα είπα την Ινδία και το Πακιστάν, ε, αφορούσε την αξιότιμη χώρα την οποία αντιπροσωπεύεται, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι, μια πυρηνική δύναμη και θέλει να επιβάλλει το μονοπόλιο ε, των, πυρηνικών όπλων σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο, δεν υπάρχει καμία απόφαση του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ που να καταδικάζει το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτο, αυτοκηρύσσεται ως παγκόσμιος ε, χωροφύλακας διότι μόνη της εκείνη θεωρεί ότι είναι ο φύλακας του διεθνούς δικαίου εκείνη θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και γι' αυτό τα είπα. Ο κύριος Μούλτσερ για ένα λεπτό. Ίσως ε, θα μπορέσει ε, το ο εμπάργο των, ο, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να ε, ισχύσει αλλά τότε οι χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα θα πληγούν περισσότερο και εάν ε, το Ιράν κλείσει τα στενά του ορμούς θα υπάρξει πραγματική πετρελαϊκή κρίση. Ξέρουμε ε, πόσο αμφιλεγόμενη ήταν η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσχημα για για την στρατιωτική επίθεση στο Ιράκ και δεν θα πρέπει κάτι τέτοιο να ισχύσει και στο Ιράν. Αλλά βέβαια ε, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και εμείς στην Ευρώπη προσπαθούμε να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής στη διαδικασία Κατζιά είναι ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική για όλους μας γιατί το πρότυπο της Ευρώπης έχει απομακρυνθεί από το πρότυπο του πολέμου και επιζητεί τις διαπραγματεύσεις στην ειρήνη και γι' αυτό ψάχνει στο Ιράν ομολόγους με τους οποίους να μπορέσει να συζητήσει γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν συμφωνούν με την τωρινή πολιτική και θα ήταν επίγον πούμε ότι πρέπει η συνεργασία πάντοτε να είναι η βάση και η προσφορά για μια μελλοντική ειρηνική συνεργασία και η διαπραγμάτευση είναι η βάση της δημοκρατίας και η φιλία ε, επιτρέπει να πλησιάσουν διάφοροι πολιτισμοί και γι' αυτό θα πρέπει να προωθηθεί μια τέτοια συζήτηση στο λαό του Ιράν. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κυρώσεις κατά του πληθυσμού, αλλά για αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν το δίκαιο και μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να συνοψίσετε ή να απαντήσετε στα διάφορα θέματα που σας ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ σημαντική και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες ε, τις παρεμβάσεις. Θα ήθελα να κάνω μία απόπειρα να συνοψίσω τα διάφορα θέματα τα οποία εκφράστηκαν εδώ και να προσπαθήσω να τα προωθήσω εντός του σκεπτικού μας για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν αρκετοί συνάδελφοι, με πρώτο και κυριότερο τον κύριο Σαλαφράγκα, είπαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τους υπολείπους και να διασφαλίσουμε ότι συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας. Όχι μόνο, αλλά συμπεριλαμβάνοντας και ε, τους, ε, τις τρεις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν ε, την Κίνα, τη Ρωσία ε, και τη ΣΥΠΑ ε, και Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία είναι οι τρει χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι χώρες κάθονται πίσω μου όταν συζητάμε με το Ιράν διότι είναι οι έξι χώρες που έχουν οριστεί ως αρμόδιες από το Συμβούλιο ασφαλεία. Αλλά Υπάρχει και ο, η Κίνα. Όταν ήμουν στην Ινδία μίλησα με τον ομόλογό μου στην Κίνα και ε, συζητήσαμε για την κατάσταση αλλά και με άλλες χώρες όπως την Ιαπωνία και την Κορέα και υπάρχει φιλοδοξία το χάσμα που θα δημιουργηθεί από τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πληρωθεί από κάποιον άλλον. Αρκετοί συνάδελφοι ανέφεραν το ρόλο της Τουρκίας. Έχω στενές επαφές με τον κύριο Νταβούτογλου για το θέμα αυτό η Τουρκία μας δίνει πολλές σημαντικές πληροφορίες, αλλά κάνει και διάλογο με το Ιράν. Είναι αυτή που ενισχύει τα μηνύματά μας, αλλά είναι και αυτή που φιλοξώνησε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων. Και νομίζω ότι συνεισφέρουν με τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν μαζί μας για το θέμα αυτό. Θα μεταβώ στη Βραζιλία αυτό το Σαββατοκύριακο για αρκετέ συζητήσει, ε, ε, μεταξύ των οποίων φυσικά θα είναι και το τι ακριβώ θα κάνουμε για το Ιράν και για ποιο λόγο. Ε, και σημειώνω όλα όσα ακούστηκαν για την ενίσχυση και τη διεύρυνση ε, του μηνύματος ε, για τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο τα κάνει και την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να συνεργαστεί για να εξεύρει την κατάλληλη λύση για το θέμα αυτό. Σε όλε τι επαφέ μα λοιπόν παγκοσμίω έχουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Φροντίζουμε να τονίσουμε ότι οι κυρώσει είναι σημαντικέ και ότι ο στόχο μα είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσω μια διτή προσέγγιση η οποία σχεδιάστηκε ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Ο δεύτερο τομέα στον οποίο θα ήθελα να σταθώ αφορά τους, το λαό του Ιράν. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε το καθεστώς του Ιράν ότι πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. παρακολουθώ τα όσα κάνουμε ώστε να μην πληχθεί η χώρα οικονομικά και να είμαστε βέβαιοι ότι οι επιπτώσεις για το λαό του Ιράν να είναι οι ελάχιστες δυνατές αλλά ταυτόχρονα να κατανοήσουν και τι ακριβώς κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί Ιρανοί πολίτες που συμφωνούν με αυτό που φιλοδοξούμε να κάνουμε και εμείς. Ε, θέλουν να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα και ε, προσπαθούμε με τα κράτη-μέλη να δούμε και τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα όσα γίνονται μέσω των κυρώσεων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοούμε τι κάνουμε και ότι εξετάζουμε και τα αποτελέσματα. Τα ε, εθνικά νομικά συστήματα προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει παράκαμψη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται για το θέμα αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι το στρατόπεδο Ασράφ έχει και Ιρανούς πολίτες. Αναφέρθηκα ε, αρκετές φορές στη σημασία που δίνουμε στην εξέβριση μιας ικανοποιητικής λύσης ε, για τους ε, κατοίκους του στρατοπέδου ΑΣΡΑΒ. Η προσωπική μου φιλοδοξία είναι να καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο να είναι ασφαλές, αλλά και να τους προσφέρουμε και ένα μέλλον. Υπάρχουν ε, συζητήσεις στα Ηνωμένα Έθνη και με τα κρατημέλη για τα θέματα της επικότητας. Υπάρχουν και τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων. Υπάρχει ο Μαρτιν Κόμπλερ, ο οποίος ανέφερα ήδη, θα είναι εδώ αύριο. Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, με τη διεθνή κοινότητα και τα κρατούμε το θέμα αυτό στις συζητήσει μας με το Ιράν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί να βρουν ένα κάποιο μέλλον, να μην παραμείνουν απλώς εκεί στο στρατόπεδο γιατί δεν έχουμε εμεί ένα σχέδιο. Ε, μπορεί να μην είναι τέλειο το σχέδιο, είναι μια συμβιβαστική λύση, αλλά εάν γίνει με το σωστό τρόπο ε, υπάρχει δυνατότητα να έχουν ένα μέλλον αυτοί οι άνθρωποι και να είναι ασφαλείς. Και όπως σας είπα αυτός είναι ο απότερος στόχος μας. Ε, τέλος υπάρχει κάτι που είπε ο κύριος Τάνοκ ε, για το θέμα του Ιράν. Εμείς είμαστε σαφείς από του θέματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουμε να πλήξουμε το λαό του Ιράν. Θέλουμε να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουμε αυτός ο λαός που έχει τόσο μεγάλη ιστορία και πολιτισμό να μπορέσει ε, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βοηθήσει το, ε, το Ιράν να σταθεί στα πόδια του. Όταν κάποιος προσυπογράφει όμως μια συνθήκη και λέει ότι δεν θα προχωρήσει με τη διασπορά πυρηνικών όπλων έχει αναλάβει μια ευθύνη και ε, πρέπει να τη σεβαστεί. Εάν δεν γίνεται σεβαστή αυτή η ευθύνη, πρέπει κάτι να γίνει. Όλα αυτά γίνονται εντό του Συμβουλίου Ασφαλεία. Το Συμβούλιο Ασφαλεία είναι υπεύθυνο και τα θέματα επιστρέφουν στο Συμβούλιο Ασφαλεία όταν υπάρχουν ε, παραβιάσει. Και από εκεί προέρχεται και η δική μου εντολή και γι' αυτό ακριβώ προσπαθεί να ε, δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε λοιπόν οι κυρώσει αυτέ να θεωρηθούν μια πολύ σημαντική συνεισφορά ώστε να προχωρήσει η άλλη πτυχή η άλλη συνιστόσα και ε, προσπαθώ μέσω και αυτή τη οδού να ζητήσω από τους Ιρανούς να απαντήσουν στην επιστολή μου, να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουν και πάλι συνομιλίες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε έξι ψηφίσματα τα οποία έχουν υποβληθεί για την λήξη της συζήτησης. Μπορώ να κλείσω τώρα τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.